το μικρόφωνο του ομιλητού. πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα δοθούν περισσότερα χρήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια και δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει και επιτήρηση από τις ευρωπαϊκές αρχές για τις δαπάνες επιτόπου. Από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να θέσουμε και το ερώτημα των στρατοπέδων που είναι αντικείμενο διαχείρισης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Είναι εξαθλειωτικές οι συνθήκες, είναι ε, πάρα πολύ ε, φορτωμένα τα στρατόπεδα και αποκαλούνται κέντρα προσωρινής υποδοχής, αλλά ε, έχουν γίνει μόνιμες δομές. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε όσους ε, θέλουν ε, να επιστρέψουν εθελοντικά. Πώς μπορούν, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και τι δυνατότητες βλέπετε να υπάρχει ε, συμβατότητα με τους όρους ε, για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ε, πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι πρόσφυγες δεν θα λαμβάνουν μόνο συμβουλές για τη δυνατότητα επιστροφής στις χώρες προελευσής τους, αλλά και πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και τις προοπτικές τους. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καλησπέρα τη συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, από το 2018 όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 36 εκατομμύρια ευρώ 30,2 για το προενταξιακό μέσο και 5,8 σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη για να αντιμετωπιστεί και το θέμα της αυξημένης παρουσίας μεταναστών και προσφύγων στη χώρα. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο προενταξιακό μέσο, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει προστασία και ε, καταλήματα για τους πρόσφυγες ε, και μετανάστες και να καλύπτει τις ανάγκες σε είδη διατροφής ε, καθώς και ρουχισμού και καταλήμματων. Πρόσβαση στο, σε ίδρυυση παραδείγματος χάρη και υπηρεσίες υγιεινής και ψυχικής υγείας και ε, υπηρεσίε προστασίας ε, και ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προστασία των παιδιών και εκπαίδευση για τα παιδιά. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια καλύπτουν και προστασία σε αυτούς οι οποίοι ε, δεν στεγάζονται στα πραγματικά καταλήματα, αλλά στο ύπεθρο δίνει υπνόσακους, σκηνές και τρόφιμα. Τμήμα των κονδύλιων αυτών ενισχύουν τις ικανότητες της Βοσνίας Ζεγοβίνης στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, αλλά είναι μικρό κομμάτι αυτής της βοήθειας που παρέχεται. Η βοήθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντικείμενο διαχείρισης από τους εταίρους μας για θέματα διεθνού, διεθνής, διεθνούς μετανάστευσης, συγκεκριμένα από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το ERC και υπάρχουν πολύ αυστηροί όροι που πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση των κονδυλίων. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και προϋπόθεση είναι η αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τη διαχείριση που γίνεται από τον κάθε εταίρο συγκεκριμένα ε, αυτή, σε αυτήν την περίπτωση από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης αλλά και σε άλλες περιπτώσεις από τη Διεθνή ε, Αρμοστία για τους Πρόσφυγες ή άλλους φορείς. Ε, επανειλημμένα τονίζουμε στις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ότι πρέπει να είναι κατάλληλα τα κέντρα υποδοχής. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδεται εγκαίρως για να τους υποστηρίξει όπου είναι απαραίτητο. Χρηματοδοτούμε αυτή τη στιγμή έξι προσωρινά κέντρα υποδοχής, όπου βρίσκουν κατάλημα πάνω από 5.200 άτομα και οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αισθητά. Πρόσφατα, το Δεκέμβριο, κοντά στο Σεράγεβο, άνοιξε ένα νέο κέντρο υποδοχής, αλλά οι συνθήκες υποδοχής δεν είναι ακόμη επαρκείς. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Τα κέντρα αυτά προσπαθούν να στεγάσουν πρόσφυγες ε, και ε, μετανάστες που δεν θα είχαν άλλες ε, ευκαιρίες. Προσπαθούμε να τηρούνται πάντοτε οι διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα. Ευχαριστώ πολύ. Δίτμα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Μήπως έχεις κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Ένα από τα προβλήματα της χρηματοδότησης για ΜΚΟ και άλλους φορείς που διοργάνωσαν το First Aid και προσπάθησαν να προσφέρουν υλικό ήταν το πόσο προβλέψουμε τι θα κάνει με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. πέστε μας και εσείς κάτι και μετά να προσθέσει. Ναι, ναι, συμφωνώ με την ε, ερώτηση και θέλω να μας πείτε περισσότερα. Μια που είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα υποδοχής, απορρόφησης, και οι πιο ευάλωτες μετανάστες θα πρέπει να ζουν στο δρόμο. Άρα συγκεκριμένα τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης αρκετή και οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή οι άρρωστοι, οι ανήλικοι, να μην μένουν στο δρόμο. Επίσης, τι γίνεται με την προστασία, γιατί επειδή υπάρχουν αυτές οι επαναποθήσεις, στην Κροατία. Όλο ένα και περισσότεροι κολλάνε εκεί ε, σε Βοσνία Ρτζεγοβίνη Και όλο ένα και περισσότερο ζητάνε άσυλο εκεί. Μόνο τρεις τελικά όμως κατάφεραν να πάρουν το, ε, το άσυλο. Άρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να θωρακίσει το σύστημα προστασίας και έτσι να υπάρχει αρκετή πρόσφαση σε κάποια διαδικασία άσυλου. Santos, you want to add something else. Ισαβέλ Σάντος, θέλεις το λόγο. Θα επανέλθω στο θέμα των πόρων και των πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει αυτή την πολιτική, να κλείνει τα σύνορά της, να πληρώνει άλλους για να φιλοξενούν τους πρόσφυγες στη χώρα τους και κατόπιν ούτε καν να ελέγχει τι επενδύει. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε εδώ και να λέμε εντάξει, ο δώμα διάζει τους καταπλησμούς και η ύπατη αρμοστή για τους πρόσφυγες διαχειρίζεται» τους καταβλισμούς ε, στέλνουμε κονδύλια και κατόπιν οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτούς τους καταβλισμούς σε εντελώς άθλιες συνθήκες. Και το ξαναλέω, απολύτως άθλιες συνθήκες. Και εμείς ελέγχουμε τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Εμείς ε, ξέρουμε αν τα χρήματα που δίνουμε, αν η συνεισφορά μας ε, είναι μια λογική συνεισφορά ή δεν είναι αν αυτή η συνεισφορά ε, διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει ένας έλεγχος ε, της χρήσης αυτών των κονδυλίων ή δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι οι άνθρωποι που κάθεται εδώ που έχουν άμεση ευθύνη γι' αυτό, αλλά όλοι θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το θέμα αυτό. Γιατί τα κονδύλια δεν είναι αστρονομικά αλλά νομίζω ότι δεν είναι και αμεληταία. Για να την χάνουν αυτές τις μεταχείρισεις στα άτομα και θα πρέπει να ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ασυνόδευτους ανηλίκους που να μένουν μαζί με ενήλικες χωρίς να έχουν καμία προστασία γυναίκες μόνες που πραγματικά είναι ανάμεικτες, είναι σε μεικτές ομάδες χωρίς ε, καμία προστασία, δεν ε, μπορούμε εμείς να έχουμε ίση για τη συνείδησή μας λέγοντας «Α, εμείς συνεισφέρουμε, δίνουμε» τόσα μεγάλα ποσά για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί για να ανακουφίσει την συνείδησή μας. Δεν αρκούν αυτά τα ποσά. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς γίνεται ο έλεγχος της διαχείρισης κονδυλίων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια και πώς ελέγχουμε τις συνθήκες ε, σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Και θα πρέπει πραγματικά εμείς να ντρεπόμαστε που έχουμε ανθρώπινα όντα στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να συνοψίσω το πώς έχει η κατάσταση. Όσον αφορά την ε, βοήθεια, είπαμε ότι έχουμε τώρα έξι κέντρα στην Βοσνία Ριζεγοβίνη. Και είπαμε για τους πιο ευάλωτους, τους ανηλίκους, τις ε, γυναίκες, τις συνόδευτες γυναίκες, οικογένειες με παιδιά, και ήταν από τα πρώτα τα οποία κάναμε πέρσι. Καταφέραμε να φτιάξουμε μια, κάποιες νέες εγκαταστάσεις στο Μπίχατς από ένα παλαιό κτίριο, τους καλύψαμε αυτές τις κατηγορίες και έτσι τα παιδιά μπορούν να πάνε σε σχολείο. Δεν είναι ιδανική κατάσταση. Τελικά αυτό είναι αρμοδιότητα κρατική. και επειδή δεν υπήρχε πέρσι η κυβέρνηση, ήταν προβληματική κατάσταση, αλλά εμεί εξασφαλίσαμε να έχουμε αρκετές κλίνες, ε, την στέγη και κυρίως κάποιους ε, να πλαισιώνουν αυτά τα πρόσωπα που κόλλησαν σε εισαγωγικά στη χώρα, μέσα στη χρονιά και ε, ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές, είχαμε συναντήσεις υψηλού επίπεδου ε, δίκαιο και της Κομισιόν τον Ιούλιο του 1999 ε, ήταν με, με, με τους υψηλότερους αξιωματούχους της χώρας. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά κέντρα διαχείρισης. Τους πιέζαμε να αλλάξουν τη στρατηγική τους για μετανάστευση και άσυλο, το οποίο είναι προϋπόθεση για τα πάντα. Όμως, Βέβαια αυτά πρέπει να γίνουν μέσω μακροπρόθεσμα. Οπότε όμω πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον κάθε έναν που βρίσκεται στη χώρα. Και κάποιοι μετανάστες που δεν θέλουν να στεγαστούν εκεί ε, στους χώρους της ε, Ένωση. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Εκείνοι όμω που θέλουν να μείνουν εκεί πάντοτε βρίσκουμε κάποια λύση παρά τις ε, διαμαρτυρίε των τοπικών κοινωνιών τη χώρα. Μην πηγαίνουμε μόνο στη Βέλγα Κλάντουσα και στον Μπίχατς, μας λένε. Και η υπόλοιπη χώρα, μονόπλευρα πάει το βάρος, οπότε βλέπετε ότι αυτό είναι ένα ε, μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Μπόρεσε η Ομοσπονδία της χώρας να μας δώσει ε, αυτές τις εγκαταστάσεις, παλιά για τον στρατό, κοντά στο Σαράγεβο και στην Τούσλα επίσης με το που αυξήθηκαν οι μετανάστες και έτσι να αποκτήσει η χώρα δυνατότητες ε, φιλοξενίας, στέγασης ε, για αυτούς που χρειάζονται. Και, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας. το πόσο θα διαχείριζε την κατάσταση η χώρα. Συγκρίνεται το με το τι γίνεται σε Σερβία και Μακεδονία. Αλλά δεν μπορεί ακόμα η Βοσνία Ζεγοβίνη να αναλάβει τη διαχείριση των μεταναστών. Οπότε εμείς ενθαρρύνουμε βαθμία να αναλάβουν ε, από τους διεθνείς οργανισμούς αυτή τη δουλειά. Και ελπίζουμε τέλη του έτους να μπορέσουν να αναλάβουν αυτά τα κέντρα υποδοχής. Να τα διαχειρίζονται. Και θα συνεχίσουμε εμείς να πιέζουμε ε, να βρεθούν κάποιες τοποθεσίες, να δημορφωθούν κατάλληλα, που να είναι βέβαια κρατική ιδιοκτησία. Γιατί φυσικά δεν μπορούμε σε ιδιωτικό χώρο να φτιάξουμε κέντρα υποδοχής. Ε, δεν είναι και το καλύτερο. Τελευταίο, ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιες πραγματικά ακατάλληλες δομές στη χώρα και στο Βούτσεκ ήταν μια παλιά χωματερή και παρά το ότι όλοι το λέγανε κοινοβούλιο, κομισιόν, οι πάντες οι αρχές σε εκείνο το μέρος, σε Μπιχάτς και Σαρακάντων, τελικά, τελικά πίστηκαν. Για μας ήταν πολύ σημαντικό επομένως ότι έκλεισε ε, αυτός ο χώρος ε, με το που ήρθε ο χειμώνα. και επίσης κατάλληλα προσπάθειες να μην ξανανοίξει με το νέο κύμα μετανάστευση στην άνοιξη αυτός ο χώρος. Ευχαριστώ πολύ. και σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, γιατί πραγματικά ήταν μια παρέμβαση πολύ κατατοπιστική και έτσι θα θέλαμε να είναι οι παρεμβάσεις. Και δίνω το λόγο κατευθείαν στην Ιζαμπέλ, Ιζαμπέλ Βίσλερ, για τις άλλες δύο ερωτήσεις που έχει θέσει το ΕΛΚ. Ξεκινώ από την ερώτηση του κυρίου Λεπόρντε Λόπες Τζιλ. Ο ύπατος εκπρόσωπο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατόπιν του ψηφίσματος για την Κούβα το RCB 9 0200 του 2019 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019 θεωρούν ότι μπορούν να αναθεωρήσουν τη συμφωνία PDCA για το πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας. Από το 2016 η Κούβα δεσμεύεται από τη συμφωνία αυτή. Παρ' όλα αυτά τα βασανιστήρια, η αστυνομική βία, οι ε, εκτοπισμοί και οι πολιτικές διώξεις καθώς και οι αυθαίρετες συλλήψεις ε, και οι ε, φυλάκιση ακτιβιστών και δημοσιογράφων και αυτών που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν σταματήσει και ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων είναι μεγαλύτερος από 300 άτομα. Βάσει των ε, όλων αυτών λοιπόν ε, θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συμφωνία αυτή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατόπιν επαλήθευσης. Δώσω το λόγο στην κυρία Κάτια Αφέλτ για την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ με ένα γενικό σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε όρους στη συμφωνία με την Κούβα όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα θυμάστε και το 1996 σε αυτό βασιζόταν η κοινή θέση. Όμως κατέστησε σαφές ότι απέτυχε η πολιτική αυτή και δεν επέφερε την αλλαγή που ελπίζαμε. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε επιρροή και σημασία στην Κούβα. Στο μεταξύ, η πρόοδο σε ορισμένου τομεί υπάρχει, στην απελευθέρωση ταξιδίων, παραδείγματο χάρη, ή στην ε, ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει ενθαρρυνθεί και τα κράτη-μέλη με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου αποφάσισαν να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση υπάρχει στη Συμφωνία για τον Πολιτικό Διάλογο και την συνεργασία, την PDCA. Μας δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Κούβα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να μας απασχολούν. Και πρώτα απ' όλα, τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, η PDCA, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επιδίωξη των στόχων μας. Και οι στόχοι αυτοί δεν έχουν αλλάξει κατά βάση. Θέλουμε καταρχήν να υποστηρίζουμε την Κούβα στις, μετα... στις μεταρρυθμίσεις της για το πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο που μπορεί να καθυστερούν αλλά κάποιες αλλαγές υπάρχουν. Δεύτερον, προώθηση δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρίτον, συνεισφορά στη βελτίωση της ζωής των κουβανών πολιτών. Όπως είπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό κομμάτι της Συμφωνίας PDCA και να σας υπενθυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2019 έγινε ο πέμπτος διάλογος με την Κούβα στις Βρυξέλλες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία επετέφθησαν οι στόχοι του διαλόγου για μια ειλικρινή συζήτηση και πραγματική συμμετοχή. Συζητήσαμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν για την Κούβα. Και οι Κουβανοί έθεσαν ορισμένα θέματα που τους απασχολούν και αυτό βέβαια είναι κομμάτι του διαλόγου μεταξύ εταίρων. Υπάρχει λοιπόν ένα φόρουμ στο οποίο μπορούμε ανοιχτά και ξεκάθαρα να συζητάμε τα σημεία στα οποία δεν συμφωνούμε. Πολλές φορές Έχουμε δηλώσει και έχουμε διευκρινίσει προς την Κούβα ότι από αυτούς αναμένεται να τηρούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές αρχές ε, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για τους πολίτες τους. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συνεχίσουμε να θίγουμε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανησυχίες, όπως πρόσφατα με την περίπτωση του Χωσέ Ντανιέλ Φέρα. Στις 23 Δεκεμβρίου μαζί με τα κράτη-μέλη κάναμε ένα διάβημα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο συνεχίζουμε να έχουμε ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Ιζαμπέλ, θέλεις κάτι να απαντήσεις? Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Έχετε τώρα το λόγο για τη δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση προέρχεται από την Τζανίνα Ματσόρσκα. Στις 20 Νοεμβρίου γιορτάσαμε την 30η επέτειο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η πρόσφατη έκθεση του Launch Countdown υπογραμμίζει ότι ένα παιδί που γεννιέται σήμερα θα βιώσει ένα κόσμο που θα είναι θερμότερος κατά 4 βαθμούς Κελσίου από ότι ο μέσος όρος στην προβιομηχανική εποχή και ε, η κλιματική αλλαγή ε, πλήττει την υγεία των παιδιών ε, και των εφήβων μέχρι τα γυρατιά. Τα παιδιά θα είναι αυτά που θα πληττούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή παγκοσμίων. Ποια είναι τα μελλοντικά μέτρα που σκοπεύει να λάβει υπηρεσία εξωτερική δράση προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική καταπολέμηση κλιματική αλλαγή για την προστασία των παιδιών και για τις μελλοντικέ γενιές. Ε, μάλιστα, ο κύριος Ντομινίκ Πόρτερ θα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ναι, δεν μπορούμε να διαψεύσουμε τα γεγονότα. Όπως είπατε παγκοσμίω, η κλιματική αλλαγή πλήττει περισσότερο τα παιδιά και ε, σίγουρα η κλιματική αλλαγή θα καθορίσει το προφίλ της υγείας των μελλοντικών γενεών. Και χτες η Γκρέτα Τούνμπερκ στον Ταβός πάντοτε ήταν εντελώς αφοπλιστικά ειλικρινής. Ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όσους κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και η έκθεση του 2019 του Lancet Countdown επίσης ε, τονίζει τι πρέπει να κάνει ο κόσμος και πού θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε αυτά που λέμε για να έχουμε, να πετύχουμε τη φιλοδοξία του Συμφωνίας των Παρισίων 1,5-2 βαθμοί τότε ε, ένα ε, παιδί ε, θα έβλεπε στα 21 του να είχε απαγορευτεί το χρήση του πετρελαίου στη Γαλλία και θα είχε φτάσει μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κλιματική δετερότητα. Όμως, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής είναι παγκόσμιες και φυσικά χρειάζεται παγκόσμια απάντηση. Η Πράσινη Συμφωνία είναι η δική μας απάντηση στις ε, προκλήσεις. Μας επιτρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να στρώσουμε το δρόμο δεν ε, ε, είναι κάτι εύκολο, αλλά ίσως ε, είναι το πιο εύκολο και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να κάνει δεν θα έχει μεγάλο αντικτυπώ, γιατί έχουμε μόνο το 9% των εκπομπών. τώρα συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν για διάφορα τμήματα της ε, Πράσινης Συμφωνίας προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια των τροφίμων, την ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα ε, και σε τοπικό και σε πολυμερές επίπεδο. Ο κύριος ε, Μπορέλ, ο υπέτος εκπρόσωπος, ε, δείχνει πρωτοφανή αποφασιστικότητα για να πιέσει, να πείσει και να βοηθήσει άλλες χώρες να αυξήσουν τις φιλοδοξίες και τις δράσεις τους έτσι ε, λοιπόν, ε, ανέλαβε αυτή την πρόκληση ε, και το συζήτησε το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για ε, τη διάσκεψη Μαδρίτης και τη Δευτέρα είπε ότι το θέμα δεν είναι απλώς να αντιμετωπίσουμε την απρόβλεπτη κρίση αυτής της στιγμής, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εντελώς προβλέψιμη κλιματική κρίση και ίσως θα πρέπει να κάνουμε πιο βιώσιμες προσπάθειες διαφορετικά αυτές οι προκλήσεις ε, στην παγκόσμια σταθερότητα θα επιδεινωθούν. Έτσι λοιπόν ε, θα έλεγα ότι θα έχουμε συμπεράσματα για την κλιματική διπλωματία και πώς συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Οι δικές μας εντολές ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι να έχουμε ύψιστη πολιτική υποστήριξη από τους Υπουργούς Εξωτερικών και αυτό θα δώσει την έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να έχουμε μια προσέγγιση στις χώρες εταίρους και να τους ζητήσουμε να κάνουν περισσότερα, πιο συγκεκριμένα και να προσφερθούμε να βοηθήσουμε. Ε, φυσικά συνεργαζόμαστε και με τους εταίρους του G20 και με τους πιο ευάλωτους εταίρους για να διδοκοποιήσουν τις προσπάθειες προ τη μέγιστη φιλοδοξία. Έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μα, οικονομική πολιτική μέχρι εμπορική πολιτική και πολλά Υπουργεία Εξωτερικών έκαναν και τη σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και επί τη ουσία και για το πώς συστηματικά θα πρέπει να καλούμε όλους τους εταίρους μας ε, να ε, ε, λαμβάνουν υπόψη την κλιματική δράση ή να αναλαμβάνουν τις ευθύνες της έλλειψής της. Ε, για πολλά χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και μέσα από τις αντιπροσωπείες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Υιοθετήσαμε κατευθυντήριες γραμμές για το ασφαλές πόσιμο νερό και για τις συνθήκες εγγενής και φυσικά αυτό αναφέρεται περισσότερο στην ευαλωτότητα των παιδιών. Επικερπίσαμε πριν δύο χρόνια τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία και την πρόθεση των δικαιωμάτων του παιδιού και αναγνωρίσαμε την ανάγκη να εντάξουμε τα δικαιώματα του παιδιού σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις πολιτικής. Ε, πέρα από τους ε, αυστηρά επικεντρωμένους τομείς στα παιδιά και αναφέρομαι σε τομείς, επενδύσεις, εμπόριο, οικονομία και άλλους. Όλα αυτά ανήκουν στην Πράσινη Συμφωνία. Και να κλείσω λέγοντας ότι αν θέλουμε να κινηθεί ο κόσμος τόσο γρήγορα όσο πρέπει, πρέπει να σκίσουμε μια ηγετική ε, στάση σήμερα ξέρουμε ότι δεν θα προκύψει από κάπου αλλού δυνάμει της ε, σημερινής γεωπολιτικής κατάστασης. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο σημείο ανταλλαγή απόψεων με την Βερνίκα Σκοβάρ από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Νόψη της μετάβασης σε Ελπάσο και Ουάσινγκτον. Διακόπτη η συσκευή για, το, για την τηλεσυνεδρίαση. a été très sur euh, cette question euh, particulièrement. Αφορά το θέμα των μεταστών στη ε, μεθόριο την Αμερικανο-Μεξικανική ε, και επίσης έχουμε και την συμμετοχή μας στην αποστολή στις Ομένες Πολιτείες. Με τον Brexit βέβαια θα την χάσουμε την συνάδελφο, αλλά θα συνεχίσει βέβαια να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ευχαριστώ και τον Μασιμιλιάνο Μασιμιλιάνο Σμερίλιο ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας της ε, Μικτής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τις άλλες αντιπροσωπείες. Οπότε ε, έχουμε από το Ελ είπαμε κοντά μας την κυρία κύριε Σκόμπαρ και έχουμε την, την επίσκεψη στο Ελβάσο και την Ουάσιγκτον. Και επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει τη συνέχεια υπήρχαν, ε, δόθηκε στα ψηφίσματα του 2010 όσον αφορά τα σύνορα Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Και σας υπενθυμίζω ότι στο ψήφισμα είχαμε πει ότι ανησυχούμε όσον αφορά την κατάσταση βάρος μεταναστών και του άσυλο ε, στα σύνορα μεξικομερικής, ιδίως όσον αφορά τους ε, ανηλίκους. Επίσης είπαμε ότι η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής είναι πάρα πολύ ακατάλληλη, ε, ιδίως από πλευρά υγειονομική. Επίσης είπαμε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν θα πρέπει να χωρίζουν τα παιδιά από τους γονείς και θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τι διεθνεί υποχρεώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΗΠΑ. Και έγιναν διάφορες επαφές και είπαμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ξεχνά αυτούς τους ε, στόχους αν είναι δυνατόν να πιέσουμε τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε και να προσέξουμε εμείς πώς διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη την μετανάστευση τι γίνεται με αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Εσκομπάρ Μεγάλη μας ικανοποίηση, σας έχουμε κοντά μας, έχετε το λόγο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. your... Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ε, που τονίζετε τη θέση σας για αυτά τα θέματα. Το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό και στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες και την απαράδεκτη μεταχείριση των μεταναστών στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Όπως αναφέρατε, το Ελπάσο βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, θα λέγαμε, όσον αφορά την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ κατά των μεταναστών. Ο Τραμπ από την αρχή είπε ξεκάθαρα ότι θα κάνει ό,τι μπορούσε για να ελέγξει τα σύνορα, όπως ο ίδιος το αποκαλεί. Αλλά θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το Ελπάσο πριν σας πω γιατί είναι τόσο επιβλαβές, επιβλαβείς οι πολιτικές του Τραμπ. Το Ελπάσο είναι μια πολύ ασφαλής κοινότητα δύο εθνοτήτων, μία από τις ασφαλέστερες στον κόσμο. Μοιραζόμαστε και τους υδάτινους σπόρους και την ατμόσφαιρα και την ιστορία και τον πολιτισμό μας και πόλεις μας είναι γέφυρες ε, μεταξύ των δύο. Υπό κάποια έννοια είμαστε ένα νέο Ellis Island. Έχουμε το άγαλμα της ελευθερίας το οποίο θεωρούμε σύμβολο της κληρονομιάς μας και ε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ε, εγώ μπορώ να σας πω ότι το σύγχρονο Ellis Island είναι αυτό το σύνορο στο Paso και θα πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε ένα κράτος μεταναστών το Ελπάσο στο Τέξας είναι από τις ασφαλέστερες πόλεις στη χώρα και βλέποντας τις στατιστικές, οι περισσότερες κοινότητες που βρίσκονται στα νότια σύνορα είναι πολύ ασφαλέστερες από τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις, από πολλές αμερικανικές πόλεις. Ακόμη και πόλεις που είναι ίδιου μεγέθους με μας. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι ασφαλείς οι κοινότητες όπου υπάρχουν μετανάστες, όχι παρά τους μετανάστες, αλλά ακριβώς λόγω των μεταναστών. Περίπου το 40% των εκλογέων μου στο Ελπάσο είναι μετανάστες, που είναι σημαντικός αριθμός. 85% του πληθυσμού μας ε, είναι ισπανικής καταγωγής και οι ρίζες τους ε, φτάνουν βαθιά στην ιστορία του Μεξικού και είναι κάτι το οποίο σεβόμαστε, τιμάμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και όταν έρχονται κάποιοι ξένοι στην κοινότητά μας, πάντοτε τους καλωσορίζουμε με ανοιχτέ αγκάλες. Και πριν από πέντε χρόνια αρχίσαμε να βλέπουμε να φτάνουν οικογένειες από κεντροαμερικανικές χώρες στο Ελπάσο. Και για να σας δώσω το γενικότερο πλαίσιο, τα προηγούμενα χρόνια συνήθως ήταν Μεξικάνοι, άνδρες μόνοι που περνούσαν ε, ε, τα σύνορα γιατί ήθελαν να μπουν στη χώρα για να δουλέψουν, για να μπορέσουν να στείλουν χρήματα στη χώρα τους, στις οικογένειές τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Ήταν οικονομικοί μετανάστες, λοιπόν, ε, ως επιτοπλίστων που ήθελαν να έρθουν, να βγάλουν χρήματα για ένα διάστημα και μετά ήθελαν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Άλλαξαν όμως τα πράγματα πριν από 5-6 χρόνια και στην δική μας ε, κοινότητα, στη δική μας πόλη και σε άλλες ε, πόλεις του, στα νότια σύνορα, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μία αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πλέον οικογένειες και οι αριθμοί στην αρχή ήταν σχετικά χαμηλοί, αλλά κατά τα τέλη του 2018 αρχίσαμε να βλέπουμε όλο και περισσότερες οικογένειες. Άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών που έρχονταν. Και Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος, πιστεύω, είναι η ρητορική του ίδιου του Προέδρου που πυροδότησε αυτή τη μαζική έξοδο γιατί ανακοίνωσε ότι θα φτιάξουμε ένα πανέμορφο, ψηλό, τεράστιο τείχο και θα κλείσουμε τους μετανάστες έξω. Πολλές οικογένειες λοιπόν από αυτές έχουν συγγενείς στις Ηνωμένε Πολιτείε και είδαν ότι ήταν η τελευταία τους ευκαιρία να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Δηλαδή τα ίδια τα λόγια του Προέδρου ε, πυροδότησε αυτή τη μαζική έξοδο από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Και υπάρχουν, πρέπει να πούμε, συνθήκες οι οποίες ε, είναι ε, φρικτές και κινητοποιούν τον κόσμο έχει αυξηθεί η βία. Οι οικονομικές συνθήκες για τους μετανάστες έχουν επιδεινωθεί και ιδιαίτερα έχουν επιδεινωθεί διότι ο πρόεδρος δεν δίνει πια βοήθεια και δεν δείχνει θετική στάση και δεν προσπαθεί να συνεργαστεί με τους ηγέτες του νοτίου ημισφαιρίου. Γιατί όταν η Αμερική δεν δίνει πλέον, ΗΠΑ δεν δίνουν πλέον βοήθεια, ε, αυξάνεται η ανασφάλεια και γι' αυτό έρχονται περισσότεροι μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν συνθήκες ε, κρέας, φτώχειας, ε, πείνας και από αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να ξεφύγουν οι πολίτες. Η κλιματική αλλαγή κάνει τη γη τους ε, μη κατοικήσιμη και πολλές ε, οικογένειες από την Κεντρική Αμερική ε, υφίστανται αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούν πια να καλλιεργήσουν τη γη τους. Άλλες οικογένειες που είχαν ζήσει επί πολλές γενιές σε αυτή την περιοχή αναγκάστηκαν να ξεσπιτωθούν γιατί έρχονται κάποιες μεγάλες εταιρείες και παίρνουν τη γη τους. Δηλαδή όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Όλα αυτά μας έφεραν στα τέλη του 2018, όπου το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ήταν προετοιμασμένο και όχι μόνο δεν ήταν προετοιμασμένο, αλλά ε, ξεκίνησε μια κρίση που είχε δημιουργηθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Το Δεκέμβριο του 2018 δύο παιδιά μεταναστών πέθαναν ε, ενώ ήταν ε, κρατούμενα ε, από τις αρχές των ΗΠΑ. Ήταν κάτι το οποίο το είδε όλος ο λαός, ήταν απάνθρωπες συνθήκες που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και πληροφορηθήκαμε ότι η ΗΠΑ η κυβέρνησή μας δηλαδή, χώριζε τα παιδιά από τις οικογένειές τους, τα άρπαζε από τις αγκαλιές της οικογένειάς τους. Μια απάνθρωπη συμπεριφορά, ε, σκληρή συμπεριφορά και εν πολύ ε, ε, ε, σημαντική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Πολλές ιστορίες φρίκης, παιδιά που υφίστανται ψυχολογικό τραύμα, τουλάχιστον 5.000 οικογένειες χωρίστηκαν από τα παιδιά τους. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 5.000 παιδιά ήρθαν στη χώρα μας με την οικογένειά τους γιατί προσπαθούσαν να ζητήσουν βοήθεια, γιατί ξέφευγαν για να φύγουν από την εξαθλίωση και αυτό που βρήκαν στις ΗΠΑ είναι μια εξαθλίωση που ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι θα ζήσουν. Η υφιστάμενη κυβέρνηση στη χώρα μας έχει κάνει μεγάλο κακό σε μια ολόκληρη γενιά παιδιών από την, τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στις οικογένειές τους. Παιδάκια που μόλις περπατούσαν ή ε, παιδάκια νεογέννητα που αποχωρίστηκαν από τη μητέρα τους. Μπορείτε να φανταστείτε τέτοιες συνθήκες σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είμαστε μια δημοκρατία, μια από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα ακολουθούσε τέτοια στάση. Και αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα από την απάνθρωπη συμπεριφορά της κυβέρνησής μας. Και έχουμε δει και πολλές άλλες απάνθρωπες πολιτικές. Παραδείγματο χάρη, μια πολιτική που ονομάζεται Πρωτόκολλο Προστασία Μεταναστών, που όχι μόνο δεν προστατεύει του μετανάστε, αντίθετα καταστρέφει τους νόμους περί Αυτή η πολιτική γιατί ξέρετε ότι για να ζητήσει κανείς ε, άσυλο πρέπει να βρίσκεται σε αμερικανικό άσυλο και ζητάει προστασία και άσυλο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και σύμφωνα με την νομοθεσία μας θα πρέπει να ακολουθήσει η σωστή διαδικασία, θα πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία να φτάσει ο ετών άσυλο στο δικαστήριο και να εξηγήσει στην κυβέρνηση γιατί ζητάει άσυλο. Η κυβέρνηση Τραμπ αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ότι όταν ζητούν άσυλο ε, ε, κάποια άτομα, άτομα που έχουν φύγει από χώρες της Κεντρικής της Αμερικής για να ξεφύγουν από τη βία και την εξαθλίωση, αυτό το οποίο τους συμβαίνει είναι ότι τους δίνουν ένα κομμάτι χαρτί, τους δίνουν ένα φύλλο χαρτί και τους στέλνουν στο Μεξικό με μια ημερομηνία για εκδίκαση. Τους στέλνουν λοιπόν στο Μεξικό σε μια χώρα που δεν ξέρουν, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν που να μείνουν δεν έχουν τρόπο να επιβιώσουν, δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους οι οικογένειες αυτές. Και ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιούργησε ένα χώρο όπου υποθάλπεται η εγκληματική δράση. Υπάρχουν περιπτώσεις απαγωγής γυναικών, ε, βίαιης σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών από την ε, Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Μεξικό. Ε, πατέρας που προσπαθούσε να βρει πάνες για το μωρό του ήταν θύμα απαγωγής. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, άτομα που εξαφανίστηκαν, είναι πλέον αγνοούμενα. Και όλα αυτά διότι η κυβέρνησή μας αρνείται να ακολουθήσει την ομοθεσία μας περί ασύλου. Και υπάρχουν και άλλες πολιτικές που θα μπορούσα να αναφέρω, πολιτικές που δημιουργήθηκαν και είναι απάνθρωπες και τραυματικές. Η βάση αυτών των πολιτικών, το κοινό στοιχείο αυτών των πολιτικών, είναι ότι είναι απάνθρωπες ε, έναντι των πλέον ευάλωτων ανθρώπων που μας χτυπούν την πόρτα ζητώντας βοήθεια. Και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η χώρα μου θα έκανε κάποια μέρα κάτι τέτοιο σε άλλα ανθρώπινα όντα. Είναι τραυματικές οι εμπειρίες. εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν, προσφέρεται ρουχισμό στους μετανάστες, ε, κουβέρτες, υπνόσακοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, το χειμώνα, να μην πεθάνουν από το κρύο. Άνθρωποι που ε, ονειρεύονταν το αμερικανικό όνειρο, οι εθελοντές που προσπαθούν να βοηθήσουν είναι πλέον εξαντλημένοι, είναι πλέον απογοητευμένοι. Ε, έχουμε δικηγόρους, ε, γενναίους δικηγόρους που προσπαθούν να υπερασπίσουν τους μετανάστες αλλά θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ασφάλεια όταν φτάνουν σε αυτές τις περιοχές που έχουν γίνει τώρα πια επικίνδυνες. Δεν μπορεί κανείς να πάει εκεί τη νύχτα. Προσπαθώντας λοιπόν οι δικηγόροι να βοηθήσουν τους πελάτες τους να έχουν μια δίκαιη δίκη, θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους τη ζωή. Επί ώρες θα μπορούσα να σας μιλάω για τις απάνθρωπες πολιτικές της κυβέρνησής μας. Να σας πω όμως ε, κάτι το οποίο είναι και το πλέον επικίνδυνο και το πιο τρομακτικό. Οι οικογένειες αυτές τώρα πλέον ε, έχουν βγει από ε, αυτά τα οποία μας παρουσιάζει η κυβέρνηση. Πολύ λίγοι δημοσιογράφοι πλέον παρουσιάζουν το τι συμβαίνει στην πράξη και χρειαζόμαστε διαφάνεια. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε αυτά τα οποία μας αποκρύπτουν. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ όχι μόνο για το ψήφισμα, αλλά και για την προσπάθειά σας να έρθετε στο Ελπάσο, γιατί η δική σας μαρτυρία θα είναι πολύτιμη, θα μπορείτε να πείτε στον υπόλοιπο κόσμο τι συμβαίνει εδώ. Και εκτός από όλες αυτές τις τραυματικές καταστάσεις, βλέποντας την απάνθρωπη συμπεριφορά προς τους ευάλωτους αυτούς ανθρώπους, τον Αύγουστο, στις 3 Αυγούστου του 19 συνέβη κάτι που πραγματικά μας ε, πλήγωσε όλους. Ένας τρομοκράτης που ήρθε στην κοινότητα τη δική μας και ομολόγησε ότι ήρθε για να σκοτώσει ε, Μεξικάνους και μετανάστες. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση έγινε διότι οι ηγέτες της χώρας μας τροφοδοτούν το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη στενομυαλιά και την ξενοφοβία. Έχουμε ένα πρόεδρο που κατά τη γνώμη μου είναι ρατσιστής. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι δεξί χέρι του Προέδρου μέσα στο Λευκό Οίκο, ο Στίβεν Μίλλερ, είναι ένας εθνικιστής και αυτοί είναι αυτοί που προωθούν την πολιτική μας για τη μετανάστευση. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν, χρησιμοποιούν ρητορική μίσους και αυτός ο λόγος ε, μίσους έχει συνέπειες. Και γνωρίζουμε, έχοντας μελετήσει την ιστορία, γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν ε, μέσα σε μια κυβέρνηση ριζώνει ο ρατσισμός. Φοβάμαι λοιπόν για τη χώρα μου. Φοβάμαι για αυτούς τους μετανάστες που είναι ευάλωτοι. Και νομίζω ότι η φετινή χρονιά, το 2020, θα είναι πραγματικά μια ε, χρονιά που θα κρίνει το τι θα συμβεί και ε, για τη χώρα μας, για τους εκλογείς μας και θα πρέπει να συνεχίζουμε να σημαίνουμε τον κόδωνα του κινδύνου για όλους ε, τους ανθρώπους στον πλανήτη. Όταν έρχονται στην πόρτα μας άνθρωποι και ζητάνε βοήθεια, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κλείσουμε την πόρτα. Και πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας αυτό κάνουν. Ευχαρίστως να ακούσω τις ερωτήσεις σας. και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι, καταπολεμώντας οποιαδήποτε ρατσιστική τάση. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Ευχαριστούμε, Βερόνικα. Να δώσω τώρα το λόγο. Στους συναδέλφους θα ξεκινήσω με τον Μασιμιλιάνο Είστε πρώτος και μετά θα δώσω το λόγο στους υπολείπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε ένα διάλογο και να συνεργαστούμε μεταξύ των διαφορών δομών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τη Βερόνικα Εσκομπάρ για τη μαρτυρία της. Είναι σκληρή. Πρόκειται για μία μαρτυρία ωστόσο που δίνει και ένα παράδειγμα. Εσείς ε, είπατε ότι το Ελπάσο είναι ένα πιθανό μοντέλο ένταξης, δείχνοντας ότι επί της ουσίας ε, μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα αν, υπάρχουν ε, δημόσιες, αν υπάρχει μια δημόσια επένδυση, αν οι μεταναστευτικές ροές δεν γίνουν ο εχθρός και αποδιοπομπαίος τράγος. Αλλά Πέρα από το Ελπάσο υπάρχει και ένα γιγάντιο και δραματικό θέμα, το θέμα των συνόρων, ολόκληρο των συνόρων. Βλέπουμε ότι εκεί καταγράφονται θάνατοι, 497 επίσημοι θάνατοι το 2019. Και επίσης υπάρχουν και τόσοι άλλοι που δεν βλέπουμε. Η βία κατά των μεταναστών, Έχουμε 600 καταγγελίες το 2019 και ξέρουμε ότι και αυτό είναι ένα μικρό μέρος ε, της πραγματικότητας. Ε, επίσης, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο, οι ανήλικοι, τα ευάλωτα άτομα. Οι συνθήκες ε, στις οποίες βρίσκονται οι ομοφιλόφιλοι που φτάνουν στα σύνορα και οι διαφυλικικές, και συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες και η έμφυλη βία που βιώνουν ε, οι άνθρωποι που παγιδεύονται και μεταξύ των συνόρων. Έχουμε από 5-8 χιλιάδες οικογένειες που έχουν χωριστεί από το 2017 όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Οι μεταναστευτικές ροές ε, φυσικά έχουν να κάνουν ε, και με ιστορικέ υποθέσεις ε, στο Μεξικό, αλλά και με ευρύτερου ε, περιοχές. Έχουμε ροές που προέρχονται από τις ε, Ονδούρες, τη Γουατεμάλα και το Μεξικό, δηλαδή αφορά όλη την περιοχή αυτό το θέμα. Όχι μόνο το Μεξικό και τις είπε. Επίσης υπάρχει και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος που δεν πρέπει να το επιτιμήσουμε και της εμπορίας ανθρώπων αυτού του business που λαμβάνει η χώρα γύρω από τα σύνορα. Και φυσικά με αυτά τα θέματα ασχολείται και η ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και εμείς ε, ως αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού θέλουμε να βοηθήσουμε εδώ στις Βρυξέλλες ε, θα έχουμε την παρουσία της αντιπροσωπείας υπό τον συντονισμό της ε, του μέλους της Γερουσίας ε, Σιτράν ε, και θα κάνουμε και συγκεκριμένο έργο. Θα συζητήσουμε το θέμα και της έμφυλης βίας. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Σκουμπάρ για τη μερτυρία σας και θέλω να θέσω τον εαυτό μας στη διάθεσή σας για να κάνουμε μια κοινή δουλειά για να προσπαθήσουμε να δώσουμε προβολή σε όσα συμβαίνουν, αλλά και συγκεκριμένε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μασιμιλιάνο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βίσλερ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από την αποστολή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευχαριστούμε για την φιλοξενία να σας τα πω τα υπόλοιπα στα γαλλικά και πάλι ε, χαίρομαι και να σας ξαναδούμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για αυτό το θέμα διότι συνήθως αλλού κοιτάμε σε χώρες που λειτουργούν διαφορετικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή χώρες που θεωρούμε φιλικές, κυρία Σκομπάρ, ε, και γιατί λέμε ε, χώρα φίλη, γιατί είναι η Αμερική. Ή γιατί αισθανόμαστε κάποια εγκύτητα και έτσι λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όμως παντού υπάρχουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παντού πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτά. Μας είπατε όλα τα προβλήματα, να μην επανέλθω στα σημεία ένα προς ένα όμως θυμάμαι όταν συντάξαμε το ψήφισμα ότι με εντυπωσίασε το πόσες έρευνες είχαν γίνει από τις Αμερικανικές αρχές, ε, ερευνητικές επιτροπές και ένα σωρό πλήρης εκθέσεις. Άρα είναι νομοθεσία. Το Αμερικανικό κράτος έχει τα μέσα του ελέγχου. Αλλά νομίζω όμως ότι μετά τις έρευνες δεν δόθηκε συνέχεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και θέλω επ' αυτού την γνώμη σας. Τι συνέπειες βλέπετε να υπάρχουν. Μα είναι επικίνδυνο. Καλά, έχουμε και το δικό μας μεταναστευτικό, το συζητήσαμε δεν ε, είμαστε πάντα περήφανοι για το τι κάνουμε εμείς στα προβλήματα που επισημαίνουμε. Όποτε, τι να κάνουμε ούτως ώστε να βοηθήσουμε την υπόθεση αυτών των ανθρώπων στη ΣΥΠΑ. Τι να κάνουμε για όλη αυτή την ε, ρητορική της καταπίεσης, της καταστολής. Τι να κάνουμε για να αντιστρέψουμε αυτό το κατά των μεταναστών ρεύμα. Και πάλι μπράβο για το έργο σας. Ευχαριστούμε Ιζαμπέλ. Ο Ντίτμαρ τώρα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Έσκομπαρ για την παρουσίαση, για την ενημέρωση. Μας περιγράψατε πως έχει η κατάσταση στα αμερικανο σύνορα. Ε, δεν είναι και τόσο διαφορετική από την κατάσταση στην Ευρώπη, όπου τα εξωτερικά σύνορα, για παράδειγμα στην Μεσόγειο, έχουμε 35.000 ασυνόδευτους ανηλίκους άντρες, γυναίκες που ρισκάρουν τη ζωή τους. Τα κέντρα υποδοχή ε, είναι πάρα πολύ γεμάτα ξεχυλίζουν. πω ε, στην έχουμε και τις νάρκες. Ε, αυτά που λέτε δεν είναι και τόσο διαφορετικά από αυτά που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Και σας ρωτώ οι Αμερικανικέ αρχές αναλαμβάνουν κάποιες στοχευμένες ενέργειες εκεί, στη Μεθόριο. Μα τι γίνεται, υπάρχει νομική βάση για αυτές τις ε, ενέργειες που κάνουν ε, έρευνες, ε, παίρνουν τα κινητά και ψάχνουν. Τι κάνουν οι αρχές, κάνουν κάτι για να μην υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοιου είδους κακοδιοίκηση και διαχείριση της ποινική δικαιοσύνης από Ονδούρα Σαλβαδόρ, ένα σωρό κόσμος που προσπαθεί να φύγει για πολλούς λόγους και ένα βασικό ε, είναι ότι είναι από τι πιο βγαίνει του κόσμου, γιατί το Μεξικό δεν θέλει να ερεθίσει τι ΗΠΑ. Τη Δευτέρα είπε ο Κάρλος Μαρτίνες ότι ο τείχος κατάπιε το τελευταίο καραβάνι στα ίδια τους πήγαν και τους κλειδώσανε κάπου αφού τους χώρισαν σε ε, ομάδες και πρόκειται να τους διώξουν, να τους απελάσουν. Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς βλέπετε το μέλλον. Ειρήνα, από το Ρήνιο. Ευχαριστώ πολύ. Βερόνικα, είναι υπέροχο που σε ξαναβλέπουμε και ευχαριστούμε για την υποδοχή σου στην Washington. Χαίρομαι που σε βλέπω τις τελευταίες μέρες της ε, θητείας μου και λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να ε, πάω στην ε, αποστολή αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο μέλλον και θα συνεχίσω να παρακολουθώ τι γίνεται με αυτές τις οικογένειες στα σύνορα που μας είπες. Από την αρχή της υπόθεσης που φτιάξαμε εκείνο το ψήφισμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνει αυτή η αποστολή, το θέμα να παραμείνει επί της τραπέζης, εδώ για μας στην Ευρώπη. Και πέρσα τη είπα ως φοιτήτρια πάρα πολύ καλά τρία χρόνια. Και πάντοτε θεωρούσα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εγγυητής της πολυμερούς πολιτικής, των δικαιωμάτων και να μην ξεχνούμε ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ήρθαν στην Αμερική είτε ως οικονομικοί μετανάστες ή ως πρόσφυγες ε, που είχαν πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και με σώκαρε πάρα πολύ όταν ε, διάβασα τα νέα αυτές από τρόπες εικόνες με τα παιδιά που τα παίρνουν στην οικογένειά τους και με αυτή την ε, καταπάτηση των δικαιωμάτων μέσα στο έδαφος των ΙΠΑ ε, εις βάρος των πιο ευάλωτων. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο το σοκ καθε αυτών των παραβιάσεων των δικαιωμάτων αλλά επίσης είναι και το σοκ ότι αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς ως δυτικοί όλο ένα και περισσότερο χάνουμε, ξεχνάμε τη διοντολογία μας, την ηθική μας και μετά μιλάμε για τα κράτη παραβάδες. Να, που όλα αυτά ισχύουν και για κάποιους στην Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που κατηγορούν. Οπότε και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί το έργο της αντιπροσωπείας Ευώσινων και ελπάσω το θέμα θα παραμείνει υποσυζήτηση και θα συνεχιστεί η πίεση προς ε, την κυβέρνηση της Αμερικής. Άρα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει η αντιπροσωπεία. Ποια θέματα θέλετε εμείς να θέσουμε. Ήδη έχω θέσει κάποιες ερωτήσεις και είτε μου απάντησαν αρνητικά, μια ξερή άρνηση ή τίποτα δεν μου είπαν. Πώς μπορούμε να έχουμε στοιχεία τα οποία να προσκομίσουμε κάποια στοιχεία που να τα δείξουμε στους Αμερικανούς. Ξέρεις κάποιες οργανώσεις ενωτών δικαιωμάτων να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους γιατί πρέπει να βρούμε επιχειρήματα τεκμηριωμένα όταν πάμε εκεί. Επίσης, ποια είναι τα προγνωστικά για φέτος, όχι για τις εκλογές, όχι δεν θέλουμε να συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά από πλευράς πολιτικής και αλλαγές που θα συμβούν φέτος. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ Σάντος. Μικρόφωνα παρακαλούμε για την ομιλήτρια. No, it's functioning. Okay. Γεια σας, χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε και ελπίζω να σας δω και πάλι σύντομα. Σας άκουσα και σκεφτόμουν ότι η έλλειψη μνήμης ε, είναι κάτι που χαρακτηρίζει Συγγνώμη, είναι κάτι που μας κάνει να χάνουμε την ανθρωπιά μας. Ξεχνάμε ότι είμαστε κι εμείς μετανάστες, πρόσφυγες στην Ευρώπη και το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η μνήμη είναι κάτι που μας ε, κάνει πραγματικά ανθρώπινους ή μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπιά μας. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις για σας. Φυσικά εδώ στην Ευρώπη διαβάζουμε διάφορες ειδήσει για το τι συμβαίνει στο Μεξικό και κοντά στα σύνορα με την εμπορία ανθρώπων. και την ε, κακοποίηση που υφίστανται οι άνθρωποι που προσπαθούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ Πολιτείες και ταυτόχρονα διαβάζουμε για όλες αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που γίνονται στα κέντρα μεταναστών. Οι συνθήκες στα κέντρα των μεταναστών είναι, σύμφωνα με τις ειδήσει που έχουμε, ότι οι συνθήκες είναι πολύ κακές. Και δίνονται όχι και τόσο λίγα χρήματα στις ιδιωτικές εταιρείες για να αιτιολογήσουν τέτοια μεταχείριση. Και αυτό έγινε πραγματική μπίζνα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ. Και εγώ έχω μια ερώτηση, Βερόνικα. Όταν μιλάμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε, πάντοτε μιλάμε για ε, τον πολυμερισμό και τώρα η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανήκει πλέον στο πολυμερέ σύστημα και πάντοτε μιλάμε για το εμπόριο, ενίοτε για το περιβάλλον, Δεν μιλάμε για τη Συμφωνία των Περσίων, όμως ποτέ, ποτέ δεν μιλάμε για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Δηλαδή το γεγονός ε, ότι δεν συμμετέχει σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Έχετε ένα θέμα στις είπα γι' αυτό δηλαδή πώς ε, γίνεται αντιληπτό το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση στο πολυμερές σύστημα σε σχέση με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες. Έχετε το λόγο. Υπάρχουν, ε, ακούσα πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες ε, και θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου. Όλες είναι εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω ομοδοποιημένες απαντήσεις. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις της Ζαμπέλ, για το ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τους μετανάστες. Και ξέρετε, υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις στο Κογκρέσο, όμως δεν υπάρχει follow-up. Και το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να μην χειροτερεύσουν τα πράγματα. Μία από τις δράσεις που αναλάβαμε πέρσι ήταν να καλέσουμε τα μέλη του Κογκρέσου να έρθουν στα σύνορα. Είχαμε πάνω από 12 αντιπροσωπείες μέλη του Κογκρέσου που ήρθαν στο Ελπάσο. Και όταν, αν δούμε τα ποσοστά, μιλάμε για το 17% των μελών του Κογκρέσου που ήρθε στο Ελπάσο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί σταματήσαμε μετά τα τέλη Ιουλίου ε, να δεχόμαστε ε, μετανάστες ε, λόγω των πυροβολισμών. Ίσως φέτος, επειδή είναι χρονιά εκλογών, είναι δύσκολο να ταξιδέψουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια περίοδου. Θα προσπαθήσουμε όμως. Όμως, τι θέλω να πω, ότι μέσω αυτής της διαδικασίας που άνοιξε τα μάτια πολλών ε, μελών, κάναμε πρόοδους για να υπάρξουν αλλαγές ε, στο Υπουργείο Ιστορικής Ασφάλειας. Όχι τεράστιες αλλαγές, αλλά κάποιες μικρές αλλαγές. Επίσης, κρατήσαμε ζωντανή την ιδέα ότι θέλουμε να ελέγχουμε την κυβέρνηση μέσω των χρημάτων που της δίνουμε δεν ε, ήταν τόσο επιτυχής ε, η πρωτοβουλία θέλαμε και ξέρετε, ενώ η Βουλή των Υπερσώπων ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, η Γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Επομένως, στο συμβασμό φαίνεται ε, πάντοτε να χάνουμε στις ενέξεις με τα χρήματα. Τώρα, τα, ο εθνικός ε, τύπος ε, δεν δίνει τόσο μεγάλη προσοχή πλέον ε, και μπορώ να σας πω μέλη του Κογκρέσου συχνά με ρωτάνε τι συμβαίνει. Εγώ ενημερώνω τους συναδέλφους και φυσικά συνεργαζόμαστε και με τις επιτροπές που ελέγχουν την κατάσταση, την Επιτροπή που, για την Εσωτερική Ασφάλεια, αλλά και άλλες επιτροπές για να ελέγχουμε την κυβέρνηση μέσω των κονδυλίων που δίνουμε θέσατε μια ερώτηση για το πώς παρουσιάζουμε το θέμα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για αυτό το διάλογο και την επίσκεψή σας ε, στην ε, Ουάσιγκτον αλλά και την επίσκεψη που θα κάνετε στο Ελπάσο και πολύ το αναφέρετε στα σχόλιά σας. Αυτό συμβαίνει παγκοσμίω. Βλέπουμε ότι αλλάζουν τα μεταναστευτικά μοντέλα και αυξάνεται γιατί υπάρχει ανατεραχή στον πλανήτη και λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω του πολέμου, λόγω της ανέχειας. Έχουμε πολλούς λόγους. Για αυτό λοιπόν είναι κοινό και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην ε, ε, χώρα καθενός, είτε πρόκειται για τη δική μου που εισαυλείται, για τη δική σας, για να βρούμε από κοινού λύση. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς οι διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές ροές, κάτι που είναι απόλυτα φυσικό. Οι άνθρωποι μετακινούνται, μετακινούνται παγκοσμίω. Αλλά ε, τότε όταν ε, δεν το συνειδητοποιούμε δημιουργούμε προβλήματα. Το Μάρτιο πήγα στην Ιορδανία με μέλη της Επιτροπής μου. Εγώ είμαι ε, στην Επιτροπή για τις Ένοπλες ε, Υπηρεσίες. Πήγα στην Ιορδανία και στη Βαγδάτη. Στην Ιορδανία πήγαμε στα σύνορα και θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σύνορα στον κόσμο. Δεν είχαν ούτε τείχος, ούτε φράχτη, ούτε μεταχειρίζονταν τους πρόσφυγες ως εγκληματίες. Και περάσαμε από ένα κέντρο από τις ζητήσαμε να το δούμε. Κάναμε εκεί μια βόλτα και οι επικεφαλής εκεί. Ε, να κάνω και μια παρένθεση στο Ελπάσο, φτάνουν χιλιάδες άνθρωποι στην κοινότητά μας. Ε, άνθρωποι κρατούνται στις, ε, στα δικά μας κέντρα για 30, 60, 90 ημέρες σε απόλυτα αξιοθρύνητες συνθήκες, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε μπάνιο για εβδομάδες, χωρίς ποιοτικά τρόφιμα ε, και ε, θα ε, πάμε λοιπόν στην Ιορδανία και τους ρωτάω πόσο χρόνο σας χρειάζεται για να επεξεργαστείτε την είσοδο των προσφύγων. Η ιδέα της επεξεργασίας είναι να συνδέσουν τους πρόσφυγες με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι να τους βγουν στη φυλακή, να τους ποινικοποιήσουν. Για αυτούς το να επεξεργαστούν την είσοδο των προσφύγων είναι να τους βρουν ένα τόπο να ζήσουν και έναν ε, τρόπο να επιβιώσουν. Πόσο χρόνο ε, πόσο χρόνος σας χρειάζεται, ρώτησα και η γυναίκα που μας ε, ξεναγούσε είπε, αντρέπομαι να σας πω, γιατί ε, μας παίρνει αρκετό χρόνο. Δύο ώρες χρειάζονται. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ είναι ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε με μετανάστες σε μια πολύ πιο πλούσια χώρα με πόρους που άλλες χώρες ε, θα επιθυμούσαν να έχουν. Κρατάμε τους μετανάστες μέχρι 90 μέρες για να τους ποινικοποιήσουμε και όχι να τους βοηθήσουμε. Επομένως, αυτή η εμπειρία στην Ιορδανία μου άνοιξε τα μάτια και μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Δεν είναι τέλεια η διαδικασία και σίγουρα δεν είναι τέλειο το περιβάλλον. Όμως ο λόγος ε, που σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα είναι γιατί θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ως μια επιμερισμένη ευθύνη και ως μια επιμερισμένη υποχρέωση, έτσι ώστε να έχουμε και κοινέ λύσεις και προκειμένου να λογοδοτούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Και ένα από τα κοινά προβλήματα φυσικά είναι η κλιματική αλλαγή δεν ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να βλέπουμε αυτές τις προκλήσεις ε, σαν ε, κουτάκια, ότι αυτό το κουτάκι είναι δικό μου, αυτή είναι η χώρα μου, μείνω μακριά, σε με μόνο μου και θα το αντιμετωπίσω. Εδώ μιλάμε για τον κόσμο και μοιραζόμαστε τέτοια προβλήματα και μπορούμε να μοιραστούμε τις ίδιες λύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος που θα πρέπει να το συζητήσουμε είναι καταρχήν να συνεχίσουμε τη συζήτηση και δεύτερον θα πρέπει να συζητήσουμε για το τι λειτουργεί και τι είναι απαράδεκτο. Τώρα, με ρωτήσατε για την παρακολούθηση ε, των δικηγόρων και των ανθρώπων που βοηθούν τους ε, μετανάστες. Προσπαθεί η κυβέρνηση να τους εκφοβήσει, τους ε, ακολουθεί, τους σταματά στα σύνορα. Τι μπορεί να κάνει το Κογκρέσο. Λοιπόν, πραγματικά αυτό ανησύχησε εμένα και τους συναδέλφους μου και στείλαμε μια σειρά επιστολών ε, βασικά για να ανοίξουμε το θέμα και να προσπαθήσουμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Χαίρομαι που το αναφέρατε γιατί θα πρέπει να επανέλθω και να δω τι συμβαίνει και τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Ήθελα να μιλήσω για το ρόλο του Μεξικού γιατί πραγματικά με ανησύχησε και με προβλημάτισε το γεγονός που το Μεξικό και συγκεκριμένα ο πρόεδρος συνεργάζεται με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με έναν τρόπο που θεωρώ ότι δεν είναι παραγωγικός. Ναι, πιστεύω ότι το Μεξικό θα πρέπει να παρακολουθεί τα δικά του σύνορα και θα πρέπει να αποτελεί σύμμαχο όμως ε, τελικά έχουν υποκύψει σε αυτό που κάνει ο Τραμπ ε, ουσιαστικά εκφοβίζει και απειλεί άλλες χώρες, απειλεί τους ε, συμμάχους και χρησιμοποιεί το εμπόριο γι' αυτό και φυσικά το Μεξικό θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Όμως, ξέρετε, μοιραζόμαστε ε, το ημισφαίριο και όλοι θα πρέπει, όλοι οι ηγέτες θα πρέπει να είναι στο τραπέζι για να βρουν λύσεις. Οι λύσεις ε, που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι λύσεις, απλώς μας οδήγησαν σε μια πιο οξία ανθρωπιστική κρίση, γιατί έχουμε μετανάστες που στέλνονται πίσω σε πολύ επικίνδυνες χώρες δηλαδή μέσω των συμφωνιών για τις ασφαλείς τρίτες χώρες. Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, αλλά οι χώρες αυτές δεν είναι ασφαλείς. Και όλοι οι συμμαχοί μας, ε, οι γειτονέ μας, φοβούνται τον Ντόναλτ Τραμπ. Επομένως, ε, πρέπει να τα αναδείξουμε όλα αυτά και πρέπει στο Κογκρέσο να δημιουργήσουμε ένα εμπόδιο για τον Ντόναλτ Τραμπ. Θα προχωρήσω και στην επόμενη ερώτηση ποιο είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει την προσωπία που θα επισκεφτείτε το Ελπάσο, τι ερωτήσεις μπορείτε να θέσετε και προβλέψεις για την πολιτική φέτος. Θα είναι δύσκολη χρονιά φέτος και θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Γιατί συμφωνώ ότι δεν θα μπούμε σε συζητήσεις ε, για την πολιτική αυτή καθ' αυτή. Αλλά επειδή πρόκειται για χρονιά εκλογών ε, για τον Πρόεδρο, και για το Κογκρέσο και για κάποια μέλη της Γερουσίας. Φοβάμαι ιδιαίτερα ότι ο πρόεδρος θα αυξήσει τη σκληρότητα προκειμένου να φανατίσει τη βάση του. Έχουμε πολλούς ψηφοφόρους στη χώρα μας που πραγματικά χαίρονται πολύ με όσα κάνει ο πρόεδρος τους μετανάστες. Είναι πραγματικά ενοχλητικό και φοβάμαι ότι τα χειρότερα δεν έχουν έλθει ακόμα. Εγώ ε, υπηρετώ και σε μια επιτροπή που αφορά τους Ισπανόφωνους και είπα ότι φέτος θα πρέπει ε, μέσω της διαδικασίας ε, θα πρέπει να πιέσουμε τους υπόλοιπους συναδελφούς να μας στηρίξουν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουμε την κυβέρνηση. γιατί μάλλον ε, έρχονται πολύ σκληρές εποχές που δεν μπορώ καν να τις φανταστώ. Φυσικά, ε, ξέρω ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να το κάνει, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κρατάς ε, όμοιρο την κυβέρνηση, είναι ακραίο και θα μπορούσε να έρθει ως μπούμεραγκ και να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε φέτος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν το όνομά του κρίνεται και είναι στο ψηφοδέλτιο. Και όταν θα έρχεται στο Ελπάσο θα έχουμε και μια μεγάλη ομάδα υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, ανθρώπων που βοηθούν ε, τους πρόσφυγες, που ε, ανοίγουν κέντρα φιλοξενίας. Θέλω να καταλάβετε ε, αυτά που αντιμετωπίζουν καθημερινά και αυτέ ε, οι συζητήσει θα σας βοηθήσουν ε, να δημιουργήσετε και τις ερωτήσεις σα, γιατί η κατάσταση αλλάζει εβδομάδα τη εβδομάδα Όταν θα έλθετε, θα έχουμε κάποιες προτάσεις για σας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να μπείτε και στην μεξικανική πλευρά, γιατί έχει νόημα να επισκεφθείτε το μέρος όπου ακριβώς βρίσκονται οι μετανάστες ε, στα σύνορα και νομίζω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να συμβεί αυτό γιατί θα είναι πολύ σημαντική συνιστόσα του ταξιδιού. Όμως, ε, καταρχήν, ε, θα γνωρίσετε όλους τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά εδώ επί τόπου, θα μπορέσετε να θέσετε διάφορες ερωτήσεις ε, και πιστέψτε με ότι θα δείτε πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Οι ιδιωτικές που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ε, πραγματικά, ε, οι συνθήκες στα κέντρα αυτά είναι πολύ άσχημες το Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλειας συνεργάζεται με έναν οργανισμό που λέγεται GSA και αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά αναθέτει όλα τα συμβόλαια εξ ονόματος του Υπουργείου Εσωτερική Ασφάλειας. Αλλά προσθέσαμε ότι υπάρχει ένα μοντέλο. Όταν το Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλειας λέει χρειαζόμαστε μια εγκατάσταση για να στεγάσουμε αυτούς τους ε, μετανάστες ε, και θέλουμε μια ιδιωτική εγκατάσταση, GSA, υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει έναν ε, διαγωνισμό έτσι ώστε πολλές εταιρείε ε, να έρθουν και να υποβάλουν προτάσεις. Βλέπουμε ότι εξακολουθούν ότι έχουν το μοντέλο να κατευθύνουν τη διαδικασία για πολύ συγκεκριμένες εταιρείε που έχουν ε, και ε, πολύ άσχημη φήμη και τους δίνουν συμβόλαια για 10 χρόνια και όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιστικό αυτό αλλά τελικά δεν λογοδοτούν και οι άνθρωποι αυτοί έτσι λοιπόν με την ομάδα μου το συζήτησα αυτό πρόσφατα για το πώς μπορούν να λογοδοτήσουν και ίσως να ξεκινήσουμε και μια έρευνα για τις πρακτικές αυτές, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα ενισχυτικό. Ναι, πραγματικά και εμείς ανησυχούμε όσο και εσείς ε, και αναζητούμε οδούς ε, έρευνας. Και τέλος, πώς ε, Αντιλαμβάνεται οι Αμερικανοί το γεγονό ότι δεν συμμετέχουμε πλέον στο Παγκόσμιο Σύμφωνο. Νομίζω ότι πολλοί Αμερικανοί δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Δεν ε, γνωρίζουν καν ότι φύγαμε. Ούτε καν ξέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα. Και δεν ε, έχει γίνει ευρύ αναφορά. Αλλά θα σας πω Και ξέρω ότι και η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, αναφέρει και τον Brexit νωρίτερα. Αυτό ο απομονωτισμός, αυτή η ιδέα ότι απλώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας μέσα στα δικά μας σύνορα και όλοι οι άλλοι να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να μας αφήσετε στην ησυχία μας. Και ε, αν δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε, δεν θα σας βοηθήσουμε ούτε εμείς. Και υπήρχε αυτή η παναχώρηση Κάποιο ανέφερε προηγουμένω ότι δεν ξέρουμε την ιστορία μα, δεν γνωρίζουμε το παρελθόν μα και δεν κατανοούμε από πού προήλθαμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, υπάρχει πολύ σημαντική έλλειψη κατανόηση τη σημασία τη δημοκρατία και του εκδημοκρατισμού. Και φυσικά αυτό συνδέεται με δύο μεγάλες προκλήσεις και με αυτό που είπα στην αρχή. Είμαστε ένας πλανήτης, ε, είμαστε ένας ε, λαός ε, κατά πολλούς τρόπους η κλιματική αλλαγή θα πλήξει εμάς όσο και εσάς. Και θα πρέπει τους συμπατριώτες μας να τους βγάλουμε από το σκεπτικό ότι μόνοι μας θα τα καταφέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι υπερβολικά μεγάλες οι προκλήσεις και οι λύσεις και οι ευκαιρίες υπάρχουν αν συνεργαστούμε. Γι' αυτό λέω ότι το 2020 θα είναι ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, γιατί αποτελεί ουσιαστικά μια μάχη για την ε, καρδιά και την ψυχή της Αμερικής. Και λέω στους πολίτες ότι πραγματικά ψηφίζουμε για τη δημοκρατία μας. Ξεχάστε τα ονόματα. Η δημοκρατία μας κρίνεται ο πλανήτης και πώς συνεργαζόμαστε. Είναι τεράστιες λοιπόν οι προκλήσεις για μας για να εγκαταλείψουμε ένα στον άλλο. Βερόνικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Με μεγάλη μας χαρά σε ξαναβλέπουμε και με μεγάλη χαρά να σε δούμε το Φεβρουάριο στην αποστολή μας. Γεια σου, γεια. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας ξαναείδα όλους. Γεια σας. Πριν, πριν ε, φύγεις να σε αποχαιρετήσω, να σε ευχαριστήσω και παρακαλώ εσύ να κατέβεις για την Προεδρία και να νικήσεις τον Τραμπ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, γεια σου. μετά από αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων και διακόπτη. Αποχαιρετά και τον Ιταλό κύριο. Μετά από αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων για την δημοκρατία και για το μέλλον του πλανήτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάμε στην επόμενη συζήτηση. Α, είχαμε πολλά σήμερα. Και πάμε τώρα στο σημείο 11 ανταλλαγή απόψεων με τους ε, βουλευτές από την Βενεζουέλα. Μιγγέλ Πιθάρο, επίτροπος του ΟΗΕ και κύριος, ε, η κυρία Μεχία, ε, επίτροπος του προγράμματος ΠΑΙΣ. Με τηλεσυνεδρίαση, με κάποιο βίντεο, υπήρχε ένα πρόβλημα με την μετάδοση στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν έχει επιληθεί για να δοκιμάσουμε να βρούμε τη λύση. Έχουμε μείνει πίσω όμως εσείς το πρόγραμμά μας. Πρώτα τον λόγο στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας με σχέσεις με την Μερκοσούρ. Ελπίζω ότι το πρόβλημα της μετάδοσης στο ίντερνετ έχει επιληθεί. <clears throat> αν δεν έχουμε την ε, εικόνα θα έχουμε ε, τον ήχο αλλά χωρίς ε, διερμηνία. Επομένως θα ακούσουμε το πρωτότυπο στα αγγλικά. Στη χειρότερη περίπτωση. Και καλά υπάρχει το χειρότερο σενάριο, μην έχουμε τίποτα. Υπάρχει το ενδιάμεσο σενάριο, μόνο με ήχο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτήν την ε, συνάντηση με το Βενεζολάνικο Κοινοβούλιο και την προσωπία μας. Ε, σας ευχαριστώ και να σας πω κάτι σύντομο. με τη σημερινή πολιτική συγκυρία στη Βενεζουέλα ε, είχαμε εξελίξεις σημαντικές τον Ιανουάριο του 2020 είχαμε ένα πραξικόπημα κοινοβουλευτικό ε, εις βάρος του ε, καθεστώτος Μαδούρο και ε, υπήρξε παρεμπόδιση του Χουάν Γουαϊδό για να αναλάβει τα ενία της χώρας. Βέβαια εδώ και πολύ καιρό υπάρχει ένα σχετικό ψήφισμα. Αυτά γίνονται μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο που ένα και γίνεται πιο ε, περίπλοκο γιατί έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή, πρόβλημα με φάρμακα, είναι οι ανάγκες που λείπουν και έχουμε 4,5 εκατομμύρια που ήδη έχουν φύγει από τη χώρα. Ε, το 94% τώρα στη χώρα ζουν στο κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και το νούμερο αυτό όλο αυξάνει. Και όπως λέγαμε το Κοινοβούλιο ε, εδώ και καιρό. Ε, ξέρει το πρόβλημα για το πόσο είναι ε, κατάσταση ανάγκες και γι' αυτό έχουμε 10 ψηφίσματα για τη Βενεζουέλα στην προηγούμενη θητεία. Αλλά για να σταθούμε λίγο στο τελευταίο ψήφισμα, αυτό το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία Ολομέλεια. Όπως αναφέρθηκε, 471 ψήφι κατά μίας και τρεις αποχές για ένα ψήφισμα υπέρ του Χουάν Γουαϊδό ως νόμιμου Προέδρου της Βουλής και προσωρινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Και είπαμε ότι επαναβάλλουμε την προσήλωσή μα στι θεμελιώδει Αρχέ, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, σύμφωνα με το ψήφισμα, καλούμε του αλλοδαπού ε, αρχηγού κρατών ε, μέσω του Ζουζέ Μπορέλ να αναβαθμίσουν την δράση της Ένωσης για να κατασταθεί η δημοκρατία και να αποκατασταθεί στην χώρα και αυτό δεν αφορά μόνο μια απλή δήλωση. Καταγγέλουμε το τρινικό καθεστώς Μαδούρο και είπαμε ότι είναι συγκρίσιμη καμπή για τη χώρα. Και θα πρέπει να στα κράτη-μέλη να αποκαταστήσουν τι πολιτικέ σχέσεις με τον Χον Βοηδό ως νόμιμο ε, πρόεδρο της χώρας. Αυτό είναι επίσης ο στόχος του ψηφίσματος, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, τονίζω, Πρόεδρε, ότι βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος Γουαϊδό στο Κοινοβούλιο. οποίο ε, θέλει να τον συναντήσει και πολλές αντιπροσωπείε ήδη το έχουν κανονίσει αυτό οι πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά πρέπει να πούμε ότι το ψήφισμα ως ψήφισμα δεν έχει ως αντικείμενο μόνο την αναγνώριση του κ. Γκουαϊντό. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Ο στόχος δεν είναι να τον αναγνωρίσουμε ως μόνο νόμιμο πρόεδρο, αλλά να ξεκινήσει μια διαδικασία δημοκρατική στη Βενεζουέλα. Θέλησα να το υπενθυμίσω αυτό γιατί ε, διεξάγουμε συζητήσεις με κάποιους που βρίσκονται επί τόπου, που αναλύουν την κατάσταση, με βουλευτέ που έχουν επισκεφθεί και γνωρίζουν την κατάσταση και δεν θα πρέπει ε, να περιγράφουμε πολύ συνοπτικά την κατάσταση σε σχέση με τον κύριο Γκουαϊντό και το ψήφισμα. Αλλά βέβαια οποιοδήποτε θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτά που λέω ελεύθερα. Θα δώσω το λόγο στον Μιγγέλ Πισαρό που είναι ε, Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Πίσαρο ε, έχει το λόγο και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Again, we, we have a... Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο μάλλον. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σας γιατί δεν σας ακούμε. Yeah, we don't hear you. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Yeah. Perhaps we have to restart the connection uh, to be Ας δοκιμάσουμε να έχουμε μια καινούργια σύνδεση μήπως λειτουργήσει. Okay. Um, we are... Can you hear? Τώρα μας ακούτε? Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. There is a problem. I don't know what. I think it's, it's from you. Έχει κάποιο πρόβλημα η σύνδεση. It's nothing. it's not uh, Are you sure that Δείτε άλλη μια φορά ότι λειτουργεί το, το μικρόφωνο σας, ότι το έχετε ανοίξει. <laughs> no.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 Θα προσπαθήσουμε τηλεφωνική σύνδεση, λέει η Πρόεδρος. Σας δίνουμε το λόγο, λοιπόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Okay. It's Congressman Pizarro uh, here as well. Sorry. So we have another phone call from from from Juan. But not the phone call from Miguel. Αυτή είναι η τηλεφωνική κλίση με τον Χουάν και όχι με τον Μιγγέλ. Έχουμε δύο συνομιλητές ταυτόχρονα. Πολύ δύσκολη θέση μας. Μιγγέλ! Έχουμε την εικόνα του Μιγγέλ και τη φωνή του Χουάν. will change. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον Χουάν Αντρές Μέχια, Επίτροπο για το σχέδιο. Μπορούμε να έχουμε τον Χουάν τώρα. No. We <laughs> <laughs>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 we will work by Νομίζω ότι θα έχουμε μόνο ήχο και όχι εικόνα. Και δεν θα έχουμε διερμηνία, αφού δεν έχουμε εικόνα. Θα συνεχίσουμε είτε αγγλικά μόνο είτε ισπανικά. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα θα μας μιλήσουν. Αγγλικά καλύτερα πιστεύω. je suis vraiment désolée mais la technique nous fait défaut. Paradoxalement, c'est avec l'Iran que nous avions Δυστυχώ η τεχνολογία δεν μα βοηθάει. Με το Ιράν τα πήγαμε καλύτερα, είχαμε καλύτερη σύνδεση. So, is Miguel Pissarro. So, Miguel, we will try to do it by phone only.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 αν έχουν ερωτήσει στα μέλη της Επιτροπής, εγώ έχω κάποια ερώτηση. Δίνω το λόγο στην Ιζαμπέλ Βίσλερ, Ιζαμπέλ Σάντος, στον Φιλ. Ιζαμπέλ Βίσλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη που παίρνω και πάλι το λόγο για το θέμα αυτό αλλά βλέπω το ψήφισμα και στο πρώτο σημείο βλέπω ότι μιλάμε για αναγνώριση, τον αναγνωρίζουμε ως πρόεδρο της Βουλής και προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλα. Ένα βασικό ερώτημα έχω σχετικά με το τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, κάτι που το θεωρώ αποτελεσματικό και που θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Και στο ψήφισμα για τις στοχευμένες κυρώσεις έναντι ε, ατόμων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για καταστολή. Θέλω να ρωτήσω αν είναι αποτελεσματικές αυτές οι ενέργειες και πώς ε, τα βλέπουν οι άνθρωποι εκεί. Ιζαμπέλ Ντοσάντος. Το ψήφισμα ασχολείται με πολλά θέματα που αφορούν τη Βενεζουέλα. Το ψήφισμα αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναγνωρίζει ότι η Εθνική Συνέλευση είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα και ο κύριος Γκουαϊντό είναι ο προσωρινός πρόεδρος. Προσωρινός πρόεδρος είναι κάποιος που επιφορτίζεται με το καθήκον να φέρει τη χώρα σε εκλογές. Και αυτό περιμένουμε. Η λέξη προσωρινός πρόεδρος δείχνει το σημειακό καθεστώς αυτού του ατόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει επάπειρο είναι μια λύση προσωρινή για τη χώρα. Η ερώτησή μου είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το διάλογο. Από αυτά που βλέπω μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ε, τέτοιες προϋποθέσεις για διάλογο και θέλω να ρωτήσω πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για να δημιουργηθούν συνθήκες για διάλογο, ώστε να επιληθεί η κατάσταση για να φτάσει η χώρα σε εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Φιλ Μπένιον. Μας είπαν ότι το καθεστώς ε, χρηματοδοτείται από τον πόλεμο και την κοκαίνη. Και είχαμε εσωτερικά αυτή τη συζήτηση αν θα είναι αποτελεσματικές οι μεμονωμένες κυρώσεις. Αλλά τι γίνεται με τις πιο γενικές κυρώσεις. Η ανησυχία εδώ είναι ότι οι πιο γενικέ κυρώσει έχουν επίπτωση στο λαό και όχι στο καθεστώς. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για το θέμα αυτό. Ποιε κυρώσει θα ήταν πιο αποτελεσματικέ ε, σε ποιου θα πρέπει να στοχεύσουμε και θα πρέπει να επικεντρώνεται στο πετρελαϊκό τομέα ή υπάρχουν ε, άλλες κυρώσεις που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε. που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το καθεστώς στο να λογικευτεί ή να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ο κύριος Σεζουρνέ. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε πολεμική. Φυσικά το ψήφισμα λέει πολλά άλλα πράγματα και προφανώς η κατάσταση εκεί είναι καταστροφική από, ανθρωπιστικό επίπεδο και φυσικά η πολιτική επίλυση του ζητήματος είναι απαραίτητη προπόθεση. Δεν θέλουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσουμε τη συζήτηση πιο πολύπλοκη. Θέλουμε περισσότερο να υποστηρίξουμε τους πολίτες, το λαό της Βενεζουέλα. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και να θέσω και μια ερώτηση στα Ισπανικά, αν συμφωνείτε. Σας ευχαριστούμε για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Μας ενδιαφέρει πολύ τι, συνέβη, τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Η πολυπλοκότητα της πολιτικής κρίσης δεν φαίνεται ξεκάθαρα, ούτε βλέπουμε ξεκάθαρα την έξοδο από την κρίση. Και από τους ε, βουλευτές ε, εδώ ε, υπήρξε μεγάλη ενθάρρυνση και μεγάλο όσο ότι βλέπουν την έξω από την κρίση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, ε, να ρωτήσω τι χρειάζεται από το εξωτερικό προκειμένου να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα. Γιατί μιλάμε πολύ για την κατάσταση, για το πλαίσιο. Όμως, ε, θα θέλαμε να μας πείτε και με διπλωματικούς όρους και με όρους ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι χρειάζεται. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Η Βενεζουέλα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε δια τα δικαιώματα των ηθαγενών, των αυτόχθονων λαών. Και είδαμε τους τελευταίους μήνες την επιδείνωση της προστασίας των αυτόχθονων λαών. Συχνά αυτό σχετίζεται με βούληση της κυβέρνησης Μαδούρο να εκμεταλλεύεται τη γη και τους πόρους όπου κατοικούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Ποια είναι η κατάλληλη εγγύηση, η καλύτερη εγγύηση σήμερα ενός πολιτικού συστήματος που θα επιτρέψει την προστασία των θαγενών. Σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, παράλληλες κυβερνήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν τους πόρους εκεί όπου βρίσκονται και συχνά παράνομα. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς από την πλευρά της Ευρώπης να εργαστούμε για τη δέους επιμέλεια, παραδείγματος χάρη των επιχειρήσεων, να εγγυώνται την ενχνευσιμότητα των πρώτων υλών ε, που ε, εκμεταλλεύονται και να εγγυηθούν ότι δεν προέρχονται από περιοχές σειράξεων. Μία τέτοια νομοθεσία από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί συχνά ζητάμε από τις χώρες της σύραξης να ρυθμίσουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά ενίοτε εμείς Είμαστε υπεύθυνοι για την τροφοδότηση αυτών των σειράξεων ε, μέσω των αγαθών που καταναλώνουμε. Έτσι λοιπόν, μια υποχρεωτική νομοθεσία για ε, τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την εχνευσιμότητα των ορεικτών που προέρχονται από περιοχές σειράξεων θα μπορούσε να βοηθήσει όποιο και αν ε, είναι το πολιτικό καθεστώς στο να επιφέρουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε σήμερα στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ.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 Ευχαριστούμε, Μιγγέλ. Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που γίνεται με αυτό τον τεχνικά δύσκολο τρόπο. Πάντως ε, παρακολουθήσαμε αυτά που μας είπες και θα είμαστε σε επαφή στο μέλλον σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Και δίνω το λόγο τώρα στην ε, Ινές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος Πιζάρο, οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, όπως περιγράφονται και από την Μισελ Πατσουλέ, είπα το εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να τα ε, παραγνωρίσουμε. Και έχουμε και εμείς ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Ακούσατε για τις ε, πρόσφατες βιοπραγίες κατά μελών της Εθνικής Συνέλευσης, ε, κατά της δημοκρατικής λειτουργίας της Εθνικής Συνέλευσης, που παραμένει το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στη Βενεζουέλα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Εμείς καταγγέλουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, κράτους δικαίου και το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Ομάδα Επαφής εξέδωσε περίπου 37 διακηρύξεις σχετικά με τις πολλαπλές ε, πτυχές της κρίσης στη Βενεζουέλα. Το Σεπτέμβριο υιοθετήσαμε τις επιπλέον κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων κατόπιν παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα μετά το θάνατο Καπτένα Κώστα και τώρα 25 ε, άτομα υφίστανται αυτές τις κυρώσεις. Δεδομένων των τελευταίων ε, εξελίξεων, τις 15 Ιανουαρίου, συνεχίζουμε στοχευμένες ε, προσωποποιημένες κυρώσεις που να μην έχουν επιπτώσεις επί του πληθυσμού που ήδη πλήττεται πάρα πολύ από τη γενικότερη κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα στην ε, Βενεζουέλα και θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο του για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υποστηρίξαμε τις πρωτοβουλίες της ομάδας της Λίμα και το τελευταίο ψήφισμα που δημιουργεί μια διερευνητική αποστολή. Η αποστολή αυτή άρχισε ήδη τη λειτουργία της και θα λειτουργήσει επί ένα έτος και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία και να προσπαθήσουμε να προάγουμε ε, την ε, λογοδοσία. Ήμασταν ως παρατηρητές στις πρόσφατες εκλογές στη Βενεζουέλα και προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτως ώστε να τηρούνται οι μηχανισμοί του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. στην κρίση στη Βενεζουέλα σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε και δεν μπορεί να λυθεί η κατάσταση χωρίς να έχουμε δίκαιες προεδρικές εκλογές. Και δεν αρκούν οι διακηρύξεις και οι κυρώσεις για την επίλυση της κρίσης. Αυτό το γνωρίζουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ενεργό ρόλο και με τη Διεθνή Ομάδα Επαφής Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη διεθνή διπλωματία να κάνει ό,τι μπορεί. Πιστεύουμε ότι ο μόνος πιθανός δρόμος είναι μια δημοκρατική μετάβαση. Αυτή τη στιγμή η διαμεσολάβηση έχει παγώσει και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στο μεταξύ είναι να δημιουργήσουμε το χώρο για να ξεκινήσει για άλλη μια φορά ο διάλογος για τη δίκαιη μετάβαση. Όπως είπε και ο κύριος Πιζάρο, γνωρίζουμε ότι η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης είναι δραματική. Παράλληλα με το πολιτικό μας έργο, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα και τα θέματα της μετανάστευσης στη γύρω περιοχή. Από το 2018 έχουμε δώσει περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ και αν συμπεριλάβουμε και τις προσπάθειες των κρατών μελών, η συνολική μας βοήθεια ανέρχεται στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, υποστηρίζουμε ενεργά ε, τις προσπάθειες αυτές στο μέλλον. Έχει γίνει η Διεθνής Διάσκεψη Αλληλεγγύης για την κρίση ε, του μεταναστευτικού. Συμφωνήσαμε ότι θα προσπαθήσουμε να υποστηρίζουμε τις τεράστιες προκλήσεις που τίθενται για την περιφέρεια με μια νέα διάσκεψη που πρέπει να λάβει χώρα μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2020. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής μαζί με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τόσο μας είπατε από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν μείνει μέχρι το τέλος αυτής της ημέρας, ε, η οποία ήταν ε, πλήρης ανταλλαγών. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ.